Έχουμε πάρει τη θέση του Συμβουλίου για, σε πρώτη ανάγνωση και τη θέση της Κομισιόν. Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του Κοινοβουλίου και υπάρχει από τη στιγμή δημοσίευσης μια προθεσμία τριών ε, μηνών για αντίρρηση σε σχέτη. Ερχόμαστε τώρα σε θέματα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτου δικαίου και δημοκρατίας